Το πρώτο σημείο λοιπόν αφορά την κατάσταση στη Συρία. Κανονικά θα είχαμε μαζί μα την Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή και είπατε εκπρόσωπο τη Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία. Με ενημέρωσαν ότι εφόσον εκείνη δεν μπόρεσε να είναι εδώ, θα δώσουμε το λόγο στην Λουσίντα Κρέιτον. Που θα μας απευθύνει το λόγο. Ενώπιον του Κοινοβουλίου. Δεν θα κάνουμε τη διαδικασία της ε, μπλε κάρτας. για σήμερα. Πρώτα θα ακούσουμε την Υπουργό Κρέιτον. Um, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρέψτε μου να σα ε, ενημερώσω εκ μέρου ε, τη ΕΥΠΑ, τη εκπροσώπου και αντιπροέδρου τη Επιτροπή Καθρινάστων, για την ε, εξολόγηση τη κατάσταση στη Συρία από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι σίγουρη ότι όλοι σήμερα μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η πολιτική λύση ε, <clears throat> σε αυτή την ε, τρομερή και σχεδόν ε, <clears throat> διετή σύγκρουση στη Συρία δεν βρίσκεται εν όψη. Η πολιτική διαδικασία που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνή κοινότητα έχουν στηρίξει με πραγματική αποφασιστικότητα, δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει αρκετά αυτή τη στιγμή. Ε, επίσης δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το καθεστώς Ασάντ έχει μετακινηθεί στην αδιαλαξία του. Όλοι είδαμε ε, το ύφος ε, του Προέδρου Ασάντ στην απαράδεκτη ομιλία του, όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς από τους εταίρους μας και από τον ε, κοινό ειδικό εκπρόσωπο Βρεχίμη. Από τη δική μας πλευρά εμείς ε, είμαστε ε, απόλυτοι, δεν υπάρχει μέλος για τον Ασάτ στο πολιτικό μέλλον, για τον Ασάτ στο πολιτικό μέλλον της Συρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασταμάτητα εργάστηκε με όλους τους εταίρους της σε διμερές, πολυμερές και ε, διαθεσμικό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα βιαστικά ζητήματα. Οι πολιτικές προσπάθειες συνεχίζονται και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε όλες τις ε, καθημερινές προσπάθειες που καταβάλλονται και στις Βρυξέλλες αλλά και ε, σε άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης και του κόσμου. Από πλευράς μας Μπορούμε να αναφερθούμε στην πιο πρόσφατη δήλωση τη ΥΠΑ εκπροσώπου σε ό,τι αφορά την ομιλία του ΑΣΑΤ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου που κάλυψε, κάλυψε μεγάλο μέρο τη προσέγγιση μα σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη Συρία. Πρέπει επίση να αναφερθούμε στην επέκταση του καθεστώτο κυρώσεων, την επίσημη αναγνώριση τη ε, Συριακή ε, Συμμαχία Επαναστατικών ε, Δυνάμεων και Δυνάμεων αντίστασης καθώς και τα ψηφίσματα ε, των Ηνωμένων Εθνών. Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το ενδεχόμενο να ε, επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις ε, για να σκεφτεί περισσότερη πίεση, πίεση στο καθεστώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να στηρίζει την αποστολή του κυρίου Μπραχήμη. Η δική του επιμονή ε, μας οδηγεί στο να του δώσουμε την, τον απαραίτητο σεβασμό. Ελπίζουμε ότι στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας ε, πλησιάζουμε προς ένα συμβιβασμό για να βοηθήσουμε τη Συρία προς το μέλλον της. Εδώ πέρα ε, παρακολουθούμε τους σύνεγγις. Ε, μια έκθεση του κυρίου Μπραχήμη που θα παρουσιάσει ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 29 Ιανουαρίου. Δεν μπορούσε να έρθει ε, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του Ιανουαρίου, αλλά θα τον έχουμε προσκαλέσει για τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατάφερε να ενισχύσει τις ενέργειες που έχουν ως στόχο την κάλυψη των προκλήσεων που αφορούν από ε, μια τεράστια ροή χιλιάδων προσφύγων ε, προς τις γειτονικές, ε, προς τις Συρία χώρες και εν μέσω ενός πολύ σκληρού χειμώνα. Συνεχίζεται και ο μεγάλος, μεγάλης κλίμακας εκτοπισμός εκατομμυρίων Συρίων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα για να στηρίξει και να βοηθήσει την, την αντίσταση ε, της ομάδας ε, αντίστασης στη Συρία και θα το εξετάσουμε αυτό το ζήτημα στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τον Ιανουάριο. Παρότι η οικονομική συνδρομή είναι τμήμα τη ε, λύση ε, μόνο, βοηθάει παρόλα αυτά σε τέτοιε προκλήσει. Από την προηγούμενη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διπλασιάσει όλε τι μορφέ συνδρομή εντό και εκτό Συρία. Ε, σήμερα πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 350 εκατομμύρια στην ανθρωπιστική βοήθεια Πάνε λοιπόν προ μακροπρόθεσμε ενέργειε ε, για την στήριξη των προσφύγων, ε, τη νεολαία ε, και του πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση χρηματοδοτεί δραστηριότητε όπω το πρόγραμμα Περιφερειακή Προστασία, προγράμματα συνδρομή ε, προ του ε, εκτοπισμένου, αλλά και βελτίωση ε, των συνθήκων ζωή για όσου έχουν καταφύγει στι γειτονικέ χώρε. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειε βεβαίω και καλύτερε δίωδοι παράδοση τη βοήθεια. Θα ήθελα ε, εδώ να αναφερθώ και να επικροτήσω τις προσπάθειες της Επιτρόπου Γεωργίαβα και του προσωπικού της. Οι προσπάθειές μας επίσης ε, στοχεύουν ε, στην επόμενη μέρα και στην μετάβαση που συμπεριλαμβάνει την οικονομική βοήθεια για την στήριξη της πολιτικής μετάβασης, τη θεσμική και οικονομική ανάκαμψη. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση προετοιμάζει προληπτικά μέτρα σε περίπτωση ενδεχόμενου περιστατικού με χημικά όπλα. Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε ε, εστιάζουμε στις γειτονικές με, με τη Συρία χώρες όπως η Ιορδανία και η Τουρκία. Και στις 4 σε όλες ε, τις ε, παρεμβάσεις μας εμείς έχουμε μια προσέγγιση με τέσσερα σκέλη, συμπεριλαμβάνουμε ε, τους πολυμερείς θεσμού όπως ο ΙΕ, τι οργανώσει, της Κοινωνία των πολιτών, αλλά και με κυβερνητικέ οργανώσεις και δομές πολιτών μαζί με την δομημένη στήριξη προς την αντιπολίτευση στη Συρία. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπροεδρεύει του Ευρωπαϊκού Ανθρωπιστικού Φόρουμ του ΟΗΕ και συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας ε, να βελτιώσουμε τις ε, διόδους ε, παράδοσης αλλά και σχεδιασμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετάσχει και στην συνδιάσκεψη δωρητών με πρωτοβουλία του γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν που θα λάβει χώρα στις 30 Ιανουαρίου. Δεν ξεχνάμε βεβαίω και την ανθρωπιστική διάσταση τη Συριακή τραγωδία που έχει εκτεληχθεί τα τελευταία δύο χρόνια και έχει οδηγήσει σε πάνω από 60.000 νεκρού, 2,5 εκατομμύρια εκτοπισμένου και 500.000 πρόσφυγε. Και δυστυχώ ε, αυτοί οι αριθμοί όλο ένα και αυξάνονται, ακόμα και την ώρα που μιλάμε. Όπως θα σας πει και στη συνέχεια η Επίτροπος Γεωργίευα, εργαζόμαστε ακούραστα κάθε μέρα για να ε, μετριάσουμε τα βάσανα του Συριακού λαού, όμως συμφωνούμε ότι μια τέτοια τραγωδία ε, δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς περαιτέρω δράση και πρωτοβουλίες. Ξέρω ότι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο πιο άμεση ε, στρατιωτική συνδρομή προ ε, την αντιπολίτευση. Όμω ε, οι απόψει δίστανται επί αυτού και υπάρχει ο κίνδυνο ενίσχυση τη σύγκρουση με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε την οδό που έχουμε χαράξει, στηρίζοντα τι προσπάθειε του κυρίου Μπραήμι βοηθώντας την αντιπολίτευση ε, και για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την τραγωδία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ και θα δώσουμε τώρα το λόγο στους ε, εκπροσώπους των ε, πολιτικών ομάδων. Καταρχήν για πέντε λεπτά εκ μέρους του ΕΛΚ ο κύριος Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρία Επίτροπε, αξιότιμε κυρίες και κύριοι. Ο τρόμος ε, που βιώνουν οι Σύριοι έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Εχθές έχασαν τη ζωή τους 90 φοιτητέ ε, που ήθελαν να δώσουν εξετάσεις. Έτσι λοιπόν αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός των νεκρών. Ακούσαμε τα στοιχεία, το πόσοι πρόσφυγες ε, υπάρχουν ε, μέσα ε, στη χώρα και εκτός αυτής. Ακούσαμε ότι έχει καταστραφεί η υποδομή, τα σπίτια. Η κατάσταση λοιπόν είναι αφόρητη. Πολλοί λένε ότι είναι πλέον θέμα χρόνου. Αργά ή γρήγορα ο Ασάντ θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα, αλλά δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Φαίνεται ότι η Ρωσία τελικά παρετείται από τη θέση που έχει λάβει στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Ρωσία. Είναι και υπόλογη απέναντι στην διεθνή κοινότητα σχετικά με τη θέση την οποία έχει λάβει. Την προηγούμενη εβδομάδα έλαβε μία σχετική συνεδρίαση στη Γενέβη και πρέπει να σας πω κύριε Πρόεδρε, δεν γνωρίζω ε, κατά πόσον στη συνεδρίαση αυτή ε, παρίσταντο και εκπρόσωποι της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις δηλώσεις που έγιναν φάνηκε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτή την εβδομάδα ο κύριος Ιμπραχήμι είναι στην Αίγυπτο και στη χώρα αυτή η κατάσταση είναι πολύ δυσάρεστη, αλλά υπάρχουν και ενδείξεις ότι θα επιδεινωθεί περαιτέρω και ότι θα υπάρξουν και άλλες ε, εκατοντάδες ε, νεκρών στη Συρία που θα προσθεθούν στις 60.000 που έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους. Οι Σύριοι υποφέρουν πάρα πολύ και φαίνεται ότι η χώρα αυτή έχει μετατραπεί σε κόλαση. Λόγω λοιπόν αυτής της ε, κατάστασης η διεθνής ε, κοινότητα πρέπει να πω ότι δεν ανταποκρίνεται στο ύψος ε, των περιστάσεων. υπήρξε ένα σενάριο, μια απειλή σχετικά με τη χρήση χημικών όπλων και υπήρξε και σχετική δήλωση του Γάλλου Πρόεδρου. Αυτή τη στιγμή όμως ε, το μόνο που γίνεται είναι απλά να καθυστερούν οι άμεσα εμπλεκόμενοι, να αγοράζουν χρόνο όπως λέμε χαρακτηριστικά. Ίσως ε, η αντιπολίτευση να θέλει και αυτή να οργανωθεί καλύτερα. Εν ώψη λοιπόν αυτής τη κατάστασης η διεθνή κοινότητα πρέπει να λάβει κάποια απόφαση. Εχθέ είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Μαλί και για όλες τις αρνητικές ε, επιπτώσεις. Η διεθνής κοινότητα λοιπόν καλείται ε, να λάβει αποφάσεις. Εχθές ε, συζητήσαμε για τη γαλλική πρωτοβουλία σχετικά με την πιθανότητα να συσταθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και νομίζω ότι η απόφαση ελήφθη σχεδόν ομόφωνα. Επίσης είναι απόλυτα σαφές κύριε Πρόεδρε ότι αυτή η ε, σύγκρουση ενέχει και μία ανθρωπιστική διάσταση και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Επίτροπο για τις προσπάθειες που καταβάλει. Οι πολίτες όμως περιμένουν από εμάς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο να δώσει απάντηση στην ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά ζητούν από εμάς να λάβουμε μέτρα που θα βάλουν τέλος στην αιματοχυσία και θα βελτιώσουν κάπως ε, την κατάσταση. η διεθνής κοινότητα, κυρίως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει επιτέλους να ε, δώσουν τέλος σε αυτόν τον ανθρώπινο πόνο. Σας ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράγκα. Εξ ονόματος Σοσιαλιστών, η συνάδελφος Δεκεζέρα έχει το λόγο για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ που δεχτήκατε να αντικαταστήσετε την κυρία Άστον. Δεν είναι εύκολο και είναι μια ιδιαίτερη αρχή το θέμα δεν είναι εύκολο ούτε και αυτό και θα ήθελα να συνεχίσω με βάση όσα είπε ο φίλος μου Σαλαφράγκα. Εμείς εδώ, οι Ευρωπαίοι, Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, πιστεύω σήμερα, έναν απολογισμό αυτή της ε, διπλωματική λύση και μια ανάλυση του τι πραγματικά συμβαίνει επί τόπου. Εμείς στηρίξαμε και συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ευρωπαϊκή θέση που ήταν όλα εκτός από μια στρατιωτική ε, επέμβαση δεδομένου του πλαισίου. Σήμερα α, και ξεκινήσαμε δε από την υπόθεση ότι, με, ότι ο χρόνος θα έπαιζε υπέρ μας, ότι ο, ο Σάντε θα υποχωρούσε και θα φεύγε. Μα δεν είναι βέβαιο όμως τελικά ότι ο χρόνος παίζει υπέρ μας. Αν κάνετε τώρα έναν απολογισμό της διπλωματικής λύσης, όταν βλέπετε και μιλούσαμε για 500.000 πρόσφυγες, ε, ε, αλλά υπάρχουν περισσότεροι, αν δείτε τους ε, αριθμούς των νεκρών, αν δείτε την Εμοσταγή τρομοκρατική επίθεση ε, κατά του Πανεπιστημίου του Αλέπου που προέρχεται στην ουσία από την Αλκάιντα. όταν βλέπετε πως σήμερα οι Ρώσοι είναι σαφώς ε, ε, έχουν πάρει στη Συρία και προσπαθούν να υπερασπιστούν τις αντιροπορικές δυνάμεις του Μπασάρ Ελασάντο, ξέρετε ότι οι Ιρανοί είναι επίσης επιτόπου. Ξέρετε πως υπάρχουν αποστολές από την Σαουδική Αραβία και από το Κατάρ. Ότι ένα σωρό κόσμος δηλαδή έχει εγκατασταθεί στη Συρία και άρα η κατάσταση έχει είναι τελικά τελείως έχει τεθεί εκτός ελέγχου ε, αναρωτιέστε ακόμα αν ο χρόνος παίζει υπέρ μας ή εναντίον μας και όταν βλέπω τις θέσεις ε, του ειδικού απεσταλμένου Μπρέγιμη, αυτό που μας δίνει τι είναι ε, ένα πλάνο που είχαμε πριν από 8 μήνες, όπου θα έχουμε μια προσωρινή κυβέρνηση και ο Μπασάρ θα έμπαινε στην άκρη. Μα δεν υπάρχουν αλλαγές στα διπλωματικά στοιχεία, ενώ αντίθετα επιτόπου δεν μπορούμε να μιλήσουμε πια για τον ελεύθερο Συριακό στρατό. Μα είναι αυτοί οι νέοι σύριοι που γνώριζα τόσο καλά και που πραγματικά θέλανε την ελευθερία τους ή πρόκειται πάλι για διείσδυση των σαλαφιστών. Και γι' αυτό θέλουμε απολογισμό. Και θέλουμε και ενδεχομένως μια απάντηση, ένα, ένα πλάνο β. Θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Γεωργίευα για το ανθρωπιστικό σας σχέδιο. Έχετε κάνει ό,τι μπορούσατε και εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να ενεργήσουμε έτσι ώστε να συνεχιστεί αυτή η δράση και να μην σταματήσει, να μην πάψει η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να συνεχιστεί και θέλω να σας θέσω το εξής απλό ερώτημα πέρα από τον απολογισμό. Τελικά, Υπάρχει μια πρωτοβουλία 145 ετών για να προσφύγουμε στο ποινικό δικαστήριο ε, κατά της, ε, του καθεστώτος της Συρίας. Τι ρόλο έπαιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Ξέρω πως είναι πρωτοβουλία των χωρών. Εσείς τι πιστεύετε. Αλλά η ουσία του προβλήματος είναι ότι εδώ δεν έχουμε στρατηγική εικόνα και, και κριτική ανάλυση του τι είναι η διπλωματική λύση. Σας ευχαριστώ Βερονίκ και εξ ονόματος ε, των φιλελευθέρων έχει το λόγο για δύο λεπτά η κυρία Σάκε. Thank you, President, Minister, Commissioner, colleagues. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι η συζήτηση ε, δεν μπορεί να γίνει εδώ για τη Συρία με την ίδια την ύπατη εκπρόσωπο, γιατί επιτέλους ε, αποφάσισε να έρθει εχθές εδώ μετά από καθυστέρηση 12 μηνών και να εκπληρώσει τα καθήκοντά της. Πιο σημαντικό όμως είναι η επιρροή που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο υπό την δική της την καθοδήγηση. Έχουμε μια χώρα που μας υπενθυμίζει πόσο πολύ μπορεί να διαρκέσει ε, μια σύγκρουση. Αυτό συνέβη και στη Ιουκοσλαβία και εκεί καθυστέρησε να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται λοιπόν ότι επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία και αυτό μας ενοχλεί. Για δύο ολόκληρα χρόνια σέρνεται η κατάσταση στη Συρία χωρίς η διεθνή κοινότητα να λαμβάνει απόφαση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ντροπή. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους ε, και εκτό από τους, ε, τους φόνους και τις καταστροφές που προκαλούνται από ανθρώπους και αναγκάζουν ανθρώπους, τους συμπολίτε τους ε, να εγκαταλείψουν την ε, χώρα τους. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το χειμώνα που επιδρώνει την κατάσταση ε, και κάτι πρέπει να γίνει. Ο Ιμπραχήμι και ο Μπογκδάνο για τη Ρωσία, εκ μέρους Ρωσίας συναντήθηκαν για να ξασυζητήσουν την κατάσταση στη Συρία. Το βασικότερο είναι ότι το αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών ήταν μηδανικό, μηδενικό όπως συνέβη και τις περισσότερες φορές. Αυτό που εντυπωσίασε ήταν η έλλειψη, η Τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα πού ήμασταν ε, κυρία Επίτροπε και κυρία Υπουργέ. Ας λάβουμε τουλάχιστον τώρα την πρωτοβουλία. Έχουμε το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι η βοήθεια πρέπει να φτάσει στους απλούς ανθρώπους. Και αυτό δεν αντιφάσκει με τις συζητήσεις που γίνονται σε πολιτικό επίπεδο να υπάρξουν οι δομές εκείνες που να επιτρέπουν στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως ε, σε τρόφιμα ε, και σε φάρμακα. Μόνο η Σουηδία, κανείς άλλος δεν λέει από τα ευρωπαϊκά κράτη ότι πρέπει ο Ασάντ να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Μα γιατί όμως πρέπει να σώσουμε τους Σύριους που πεινάνε, κρυώνουν, ε, είναι στριμωγμένοι ανάμεσα σε ένα δικτατορικό καθεστώς και σε ένα, στους ακραίους ε, ε, παναστάτες. Και δυστυχώς είμαστε μακράν ακόμα από το να δράσουμε όπως το απαιτούν οι περιστάσεις. Σα ευχαριστώ εξ ονόματο των Πρασίνων και για τρία λεπτά έχει το λόγο η συνάδελφο Ελένα Φλότχα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τελευταία φορά που μιλήσαμε για τη Συρία ήταν στις 12 Δεκεμβρίου στις 4 ε, το απόγευμα με την κυρία Μάλστρομ και αναφέραμε το μακάβριο αυτό σενάριο, το προβλέψαμε και δυστυχώς ένα μήνα μετά ε, έχει πραγματοποιηθεί. Εγώ πιστεύω πραγματικά, κυρία Υπουργέ, πω δεν πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την πορεία. Σίγουρα το να διατηρήσουμε την ίδια πορεία θα σημάνει το να υλοποιηθούν και άλλε μακάβριε προβλέψει. Πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Σε αυτό είναι βέβαιο και το λέω και για την ανθρωπιστική βοήθεια που δικαίω είπαμε ότι είναι σημαντική γιατί αποτελεί το 53% τη παγκόσμια βοήθεια. Αλλά αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια καταρχήν είναι πολύ άσχημα κατανεμημένη όσον αφορά τη διμερή ευρωπαϊκή βοήθεια. Γιατί η Μεγάλη Βρετανία μόνη τη δίνει σχεδόν το μισό τη διμερού ευρωπαϊκή βοήθεια αλλά έχουμε προβλήματα διοχέτευσης, ε, διότι αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια περνά τελικά από ε, την, ε, το Συριακή Ερυθράη που μένει υπό τις επιταγές του καθεστώτος. Πώς ένα καθεστώς που συστηματικά βομβαρδίζει τους φούρνους για να προκαλέσει τον λοιμό, πώς μπορεί να οργανώσει με ισότητα και όχι πολιτικό τρόπο την ανθρωπιστική βοήθεια την οποία εμείς στέλνουμε. Και μάλιστα έχουμε πολύ σημαντικές καταγγελίες από διάφορες κοινότητες και από τους πληθυσμούς που δεν φτάνει σε αυτούς η ανθρωπιστική μας βοήθεια. Περιμένω λοιπόν στις επόμενες δύο μέρες, επειδή θα αφιερωθεί μια συνεδρία σε αυτή την υπόθεση, η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί πραγματικά ε, αποτελεσματικούς τρόπους ώστε να φτάνει στον προορισμό της ανθρωπιστική βοήθεια. Και έπειτα, βρίσκουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε τονίσει στις 12 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, για να έρθει κανείς ο Σύριος στην Ευρώπη πρέπει να περάσει από τους περασματάριδες, από τέτοια δίκτυα και ακόμα χειρότερα να αγοράσει και ψεύτικα πλαστά διαβατήρια. Γιατί με συριακό διαβατήριο δεν μπορεί κανεί να φτάσει εδώ νομίμω και να ζητήσει έστω και προσωρινή προστασία στην Ευρώπη. Και όπω το είπε σωστά η Human Rights Watch, είναι λαχείο. Λαχείο είναι ποιο θα επιζήσει. Και μόνο οι οικογένειε οι οποίε είναι πολύ πλούσιε τα έχουν καταφέρει. Δύο οικογένειες χρειάστηκε να αγοράσουν πλαστά διαβατήρια για να φτάσουν στην επικράτεια την Ευρωπαϊκή. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Πολωνία. Μα πότε θα ξεκινήσει ένα σχέδιο προσωρινή υποδοχή. Έχουμε οδηγία. Οδηγία για την προσωρινή προστασία. Είναι πλέον επίγον να κινητοποιηθεί. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να διατηρήσουμε την ίδια πορεία όσον αφορά το εμπάργο για τα όπλα. Γιατί αυτό προκαλεί το αποτέλεσμα το οποίο φοβόμαστε. Δηλαδή, οι αντικαθεστοτικοί βρίσκουν τα όπλα στι χώρε του κόλπου. Και άρα ο κίνδυνο ισλαμοποίηση που ορισμένοι προτείνουν για να αρνηθούν την πρόσβαση στα όπλα τελικά έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μα είναι τελείω παράδοξο αυτό. Αναμένω λοιπόν από το Συμβούλιο τη 31 η Ιανουαρίου να εγγύψει σε αυτό το θέμα, γιατί είμαστε αντιπαραγωγικοί απόλυτα. Και τέλος, για να κλείσω, πιστεύω πως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τα όσα συμβαίνουν στην Τουρκία και τι διαπραγματεύσεις με το ΠΚΚ. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ ευάλωτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να, βάλει, να καταβάλει όλες τις, τις προσπάθειες για να επιτύχει. Μπορεί να έχει περιφερειακές επιπτώσεις μέσω του του ντόμινο που θα είναι πολύ καθοριστικές για ολόκληρη την περιφέρεια. Ευχαριστώ. Τώρα, στο όνομα των συντηρητικών, ο Δόκτωρ Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι αυτή η σύγκρουση συνεχίζεται μετά από δύο χρόνια με, το, τέτοια, με τόσους ε, νεκρούς. Μόλις χθε μάλιστα 87 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια βομβιστική επίθεση στο Χαλέπι, στο Πανεπιστήμιο. Και βλέπουμε ότι είναι γνωστή η ιστορία όπου ο καθένας ε, κατηγορεί τον αντίπαλό του. Όμως ε, αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι και, και οι δύο πλευρές πλέον κατηγορούνται για, για ακρότητες. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ε, ένα είναι το σίγουρο ότι είναι απολύτως αναγκαίο ο πρόεδρο ε, Ασάντ να εκδιωχθεί το ζωμότερο δυνατόν γιατί έχει χάσει όλη την εξοπιστία του και το καθεξή. Ε, συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο κατά του πολιτών του και είναι έμεσα ή άμεσα υπεύθυνο για τον θάνατο 60.000 πολιτών. Η Χέσβολα ε, έχουμε μάθει τώρα ότι κινητοποιεί οι πολεμιστές ενώ ο Ασάντ προετοιμάζει την υποχώρησή του. Οποιαδήποτε απόφαση να παραμείνει όμως στην εξουσία θα ήταν εντελώς απαράδεκτη για τη Δύση. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λήξει αυτή η ιστορία. Θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο αν η Ρωσία ε, σταματήσει να μπλοκάρει επιτέλους τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και έχουν εμποδίσει έτσι και το, ε, τις διαδικασίες ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Λάξαρ Μπραχήμι πρόσφατα είπε ότι η Ρωσία είναι όσο αποφασισμένη είναι και η να σταματήσει αυτή η σύγκρουση και ότι αλλά θέλουμε η Ρωσία να λάβει δράση, όχι μόνο να μείνει στα λόγια. Ε, και το διακύβευμα εδώ είναι η επιτυχία του ειρηνευτικού προγράμματος. Ε, πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε ε, επιτέλους για να βοηθήσουμε το Συριακό λαό να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ από ε, την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, ο κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2013. Ε, ναι, το 2013 λοιπόν έχουμε αυτή την Real Politik και πλέον έχουμε δύο επιλογές. Ε, ένα, όλες οι στρατιωτικές ε, δυνάμεις ε, κατευθύνονται για να σταματήσουν τον Ασάντ και για να σταματήσει ο εμφύλιος ο πόλεμος και η καταστροφή των υποδομών της Συρίας και την ανθρωπιστική καταστροφή ε, τεραστίων διαστάσεων. Και να μην ξεχνάμε την αστάθεια και στις γειτονικές χώρες της Συρίας. Δεύτερη επιλογή θα έχουμε το τέλος ε, του, του πολέμου, του εμφύλου πολέμου στη Συρία, που θα είναι πλέον βασική προτεραιότητα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, με όλα τις, ε, να για το Συριακό καθεστώς. Ε, ελπίζω και το Συμβούλιο να ακούσει αυτή τη θέση μου, γιατί πλέον πρέπει το, το, ε, το βασικό να είναι το εσωτερικό της Συρίας και όχι το εξωτερικό. Δεν ακούσαμε ποτέ το Συμβούλιο να ε, λάβει θέση σε αυτό. Σε ό,τι αφορά την εθνική συμφιλίωση την, ε, και την, ε, τον τερματισμό αυτής της κατάστασης. Πρέπει να δείτε και τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό και μένουμε σε αυτό το, ζήτημα της ρεάλ πολιτικού που πλέον γίνεται άσχετο. Εγώ βέβαια ξέρω ότι είμαι και σκεπτικιστής. Ευχαριστούμε κύριε Μπέλτερ. Το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Μαρίζα Ματίας, εξ ονόματος της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Εμείς λάβαμε πληροφορίες αυτή τη βδομάδα μέσω του απεσταλμένου μας στα Ηνωμένα Έθνη ότι φέτος μπορεί να πεθάνουν 100.000 άνθρωποι στη Συρία. Μιλάμε για τους ε, χιλιάδες χιλιάδων πρόσφυγες και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει πόσες ακόμα χιλιάδες πρόσφυγες ε, θα υπάρξουν. Είναι μια δραματική κατάσταση, αλλά αυτό που είναι ακόμη πιο ανησυχητικό είναι όμως η αποτυχία της κοινωνίας των εθνών, της διεθνούς κοινότητας που δεν μπόρεσε να παρέμβει στην κατάσταση αυτή μεταξύ αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση ωστόσο στη Συρία συνεχίζει να επιδεινώνεται και κοστίζει το θάνατο χιλιάδες ε, αθών πολιτών. Αυτή η κατάσταση ε, οφείλεται στο αντιδημοκρατικό και βίο αιμοσταγές ε, καθεστώς του Ασάντ έχουν, υπάρχουν και εσωτερικές ομάδες οι οποίες όμως διευθύνονται από το εξωτερικό. οι κινήσεις των πολιτών έχουν διαλυθεί ανέκαθεν. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή η Συρία δεν είναι μόνο κατεστραμμένη από την εσωτερικό εμφύλιο πόλεμο, αλλά και από την εξωτερική, τις εξωτερικές παρεμβάσεις και γι' αυτό πρέπει να ζητήσουμε τις ευθύνες των διεθνών οργανισμών. Ωστόσο, δεν μπορούν οι δικές μας διαμάχες να επικρατήσουν τις ανάγκες ειρήνης μέσα στη Συρία. Πρέπει τελειώσει αυτός ο πόλεμος μια και διαπαντός. Ε, γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τη δική της πολιτική υπέρ της δημοκρατίας και της, Συρίας, και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή με πολιτικές που και δεν θα πρέπει να έχει καμία σχέση με τις παρεμβατικές πολιτικές του αραβικού κόσμου. Μόλις, όχι μόνο δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να δούμε και τι επιπτώσεις θα έχει περιφερειακά. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να σταματήσει ο πόλεμος και η ανθρωπιστική καταστροφή πρώτα. Σας ευχαριστώ. 1,5 λεπτό. Ο συνάδελφος Φίλιπ Κλάης. Εξ ονόματος των μία γεγραμμένα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλο ένα και περισσότερο καθίσταται ε, ε, η θέση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την Αραβική Άνοιξη και πόσο λανθασμένη ήταν αυτή η θέση. Υπήρξε λοιπόν ε, αυτή η αθωότητα, η αφέλεια ε, που φτάνει στα, στα όρια της ε, ιδεολογικής ε, αν θέλετε και τώρα βλέπουμε ότι η δικτατορία έχει αντικατασταθεί από χειρότερες δικτατορίες ε, και από την δικτατορία της Σαρία. Ε, φαίνεται λοιπόν Είδαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 500 δισεκατομμύρια ε, στους ε, αδελφού μουσουλμάνους της Αιγύπτου και είναι απίστευτο αυτό το γεγονός. Το ίδιο σενάριο λοιπόν θα επανεληφθεί και εδώ. Θα ήθελα να τονίσω βεβαίω ότι οι ακρότητες ε, του καθεστώτος ε, Ασάντ βεβαίω και θα πρέπει να καταδικαστούν και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι στη διαθεσή μα για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η Αλκάιντα ή ομάδες που συνδέονται με την Αλκάιντα να ε, βρουν έδαφος να προσφορήσουν στην Συρία. Το καθεστώς του δεν έχει πλέον μόνο το, το μονοπόλιο ε, στις ακρότητες ε, και τμήμα των ε, ομάδων των αντικαθεστωτικών έχει προσφύγει σε ακρότητες καταφύγει μάλλον σε ακρότητες και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κλάις για την παρέμβασή σας. Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν ε, αυτού του γύρου των ομιλητών εκ μέρου των ομάδων. Περνάμε στο τελευταίο τμήμα της ε, συζήτησης. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την Επίτροπο, την κυρία Γεωργίεβα. Ε, αρκετοί συνάδελφοι <clears throat> ε, σας ε, ευχαρίστησαν για τις ε, υπηρεσίες σας. Θα λάβετε λοιπόν τώρα το λόγο και μετά θα λάβει το λόγο η ε, Υπουργός ε, κυρία Κρέτον η οποία εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως την υπατή εκπρόσωπο. Κυρία Γεωργίευα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να δούμε προς τα που κατευθύνεται η ανθρωπιστική κρίση στη Συρία. Ε, από το κακό στο χειρότερο και έπονται ακόμα πραγματικά τα χειρότερα. Τις τελευταίες εβδομάδες ε, είδαμε μια ουσιαστική επιδείνωση της κατάστασης ε, στη Συρία. Και αυτό οφείλεται σε τρεις παράγοντες Πρώτον, στο ότι είχαμε πιο σκληρές μάχες. Δεύτερον, οι οικονομικές ε, συνθήκες ε, πλέον μπορούν να χαρακτηριστούν ε, καταστροφικές. Και τρίτον, ήρθε πλέον ο χειμώνας και δυστυχώς εφέτος ο χειμώνας είναι πολύ δρυμής ε, και ε, πλήττει τους ανθρώπους ε, με μεγάλη δρυμύτητα. Όσον αφορά λοιπόν το πρώτο στοιχείο, τις σκληρότερες μάχες, σας είπα είναι πολύ πιο σκληρές και όχι μόνο διαπράττονται ομότητες, αλλά το καθεστώς ασάντε είναι εκείνο το οποίο φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Ισχύει αυτό, αλλά πρέπει να πούμε ότι φρικαλαιότητες διαπράττονται και από την άλλη πλευρά. Έτσι λοιπόν η, η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεύτερον, αυτό που τώρα ε, πλήττει τους ανθρώπους και προστίθενται ε, είναι οι παράγοντες όπως αύξηση του πετρελαίου και τη τιμή των τροφίμων. Υπάρχει έλλειψη τροφίμων σε ε, χώρους όπως το Χαλέπι, στο Εγκλίπ, στη Χαμά, στη Χόλμς, σε, πόλεις όπου έχουμε σκληρές μάχες, εκεί πλέον υπάρχει και έλλειψη τροφίμων. Γι' αυτό λοιπόν ε, το κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσφέρουμε τη βοήθεια στους ανθρώπους. Και θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως ε, στα σχόλια της κυρίας Πλότρε. Ε, δηλαδή για το πώς ακριβώς ε, λειτουργεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία. Από την ε, πρώτη μέρα, από τις πρώτες μέρες που ξέσπασε ο πόλεμος, εμείς εμπλακήκαμε με τρεις τρόπους. Πρώτον, ήμασταν εκείνοι που δώσαμε τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια και επίσης προσφέραμε και ανθρωπιστική βοήθεια και στήριξη μέσα από το φόρουμ που συναντήθηκε τρεις φορές και μέσα από συναντήσεις και με την αντιπολίτευση για να μπορέσουμε να τους πείσουμε για την εφαρμογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην πεθαίνουν και αυτό να οφείλεται πολλές φορές στο ότι μερικοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η νομοθεσία υπάρχουν αυτοί οι διεθνείς νόμοι. Επειδή λοιπόν εμείς ε, εμπλακήκαμε, ενεπλάκημε αν θέλετε, γι' αυτό βοηθήσαμε τους ε, Σύριους πολλούς από αυτούς να μετακινηθούν. Ε, στην αρχή ο Ασάντ επέτρεπε να δράσει στη Συρία μόνο ο Ερυθρός Σταυρός. Εμείς όμως ε, μπορέσαμε να λειτουργούν μέσα στη Συρία πολλές ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Επτά εξ αυτών είναι πλέον ευρωπαϊκές. Πάνω από 19 φορείς ε, της κοινωνίας των πολιτών πλέον μπορούν να προσφέρουν την ανθρωπιστική βοήθεια επιπρόσθετα στον Συριακό Ερυθρό Σταυρό. Ο Ασάντ ήθελε ο Συριακός Ερυθρός Σταυρός να είναι ε, η Μισέλινος μάλλον να είναι η, ο μόνος φορές που θα προσέφερε βοήθεια. Εμείς ε, και αναφέρθηκαν τα σχετικά στοιχεία. Προσφέραμε, όπως σας είπα, οικονομική βοήθεια, αλλά προσφέραμε και κάποιο μεγαλύτερο χώρο για να λειτουργήσουν αυτοί που ασχολούνται με την παροχή ανθρωπιστική βοήθεια. Είχαμε πολλές συναντήσεις, ε, μία εξ αυτών στο Κάιρο και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μέσα στη Συρία, αλλά να βοηθήσουμε και τους πρόσφυγες, των οποίων αριθμό αυξάνεται συνεχώς. Εγώ έχω επισκεφτεί την περιοχή δύο φορές. Ε, πραγματικά ραγίζει η καρδιά σου ε, με το να βλέπεις αυτά που συμβαίνουν. Μίλησα με μια νέα κοπέλα πρόσφυγα στην Ιορδανία, που δεν έχει πάει στο σχολείο τα τελευταία δύο χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε μόνο αυτούς που χάνουν τη ζωή τους, αλλά και αυτούς που καταστρέφεται η ζωή τους. Έχει καταρρεύσει το εκπαιδευτικό σύστημα, ε, πάρα πολλά σχολεία τώρα πλέον είναι ε, καταλήματα για εσωτερικά εκτοπιστέντες. Ε, οι τραυματίες πολλές φορές παραμένουν αβοήθητοι, αλλά και άλλα οι εμβολιασμοί και αυτοί πλέον δεν υφίστανται. Πράγματι υπάρχει οξία ανθρωπιστική κρίση και είναι καθοριστική σημασία το να δουλέψουμε σκληρά για να ε, δοθεί τέλος σε αυτή την κρίση και αυτό δεν είναι μόνο απόφαση αυτών που ασχολούνται με ανθρωπιστικά αλλά κυρίως αυτών που ασχολούνται με την πολιτική. Μερικοί μίλησαν για την δυνατότητα παρέμβασης. Εδώ θέλω να σας πω το εξή. Η Συρία δεν είναι Λιβύη, η στρατιωτική παρέμβαση δεν είναι εύκολη, είναι πολύ πιο καλά εξοπλισμένη διχασμένη Συρία. Μίλησα με ανθρώπους επιτόπου και πολλοί είπαν ότι αν υπάρξει στρατιωτική παρέμβαση ε, απ' έξω θα χρησιμοποιηθούν πράγματι από το καθεστώς χημικά όπλα και άρα το αποτέλεσμα θα είναι πολύ χειρότερο. Κατόπιν τούτου η στρατιωτική παρέμβαση δεν θα βελτιώσει την κατάσταση. Πολιτική θα πρέπει να είναι η λύση που θα αναζητήσουμε όλοι να υψώσουμε τη φωνή μας και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι εμείς ε, επίσης ε, θελήσαμε να ε, επισημάνουμε το πρόβλημα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Γενικός Γραμματέας στις 30 Ιανουαρίου βοήθησε ώστε να υπάρξει αυτή η συνάντηση σχετικά με το πρόβλημα διότι πράγματι η χρηματοδότηση είναι τεράστια και δεν μπορούμε εμείς να την καλέψουμε. Ε, εκτός από εμάς ε, υπάρχουν και άλλες και άλλοι που βοήθησαν βέβαια τους ε, Σύριους. Εμείς ε, δύο φορές δραστηριοποιήσαμε τον μηχανισμό μας ε, πολιτικής προστασίας. Επίσης βοήθεια προσφέρεται από την Τουρκία και την Ιορδανία και αν τους το ξαναπεί κανείς θα ξαναπροσφέρουν βοήθεια. Πάντως πρέπει να υπάρχει αυτή η παρέμβαση διότι δυστυχώς η πολιτική λύση που είναι η μόνη λύση ακόμα δεν διαφαίνεται. Και φοβάμαι ότι αυτό θα συνεπάρξει ακόμα μεγαλύτερο πόνο για εκατομμύρια Συρίων και ο κίνδυνος να μετακυλιστεί η κρίση σε όλη τη γειτονική περιοχή. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω όλους σας εδώ στο Κοινοβούλιο ότι η ανθρωπιστική ομάδα της Επιτροπής έχει βοηθήσει ανθρώπους να μην πεθάνουν ε, από την ομάδα της ανθρωπιστικής βοήθειας 15 πέτραν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν Πραγματικά ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ. Ε, θέλουμε η Ευρώπη να δείξει τη στράτευση της ε, για να μην υποφέρουν αυτό οι άνθρωποι και το κάνουμε αυτό με όσο περισσότερα μέσα μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Επίτροπο. Τώρα να δώσουμε το λόγο στην Υπουργό Κρέιτον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα... Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τις ιδιαίτερα επικοδομητικές παρεμβάσεις τους. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και συμμεριζόμαστε τον βαθύ προβληματισμό ε, και κατανοούμε το επίγον της κατάστασης ό,τι αφορά την επίλυση αυτής της τρομακτικής ε, ε, ιστορίας που εκτελείται αυτή τη στιγμή στη Συρία, όπως ανέφερε και η Επίτροπος. Για να γίνει αυτό απαιτείται αποφασιστικότητα και συνεργασία όλων, μεταξύ όλων των θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας για να καταλήξουμε κάποια στιγμή σε μια πολιτική λύση, όπως είπε και η Επίτροπος. Στις παρατηρήσεις μου ήθελα να απαντήσω μόνο σε κάποια από τα ζητήματα που έχουν θυγεί και ζητώ συγγνώμη αν ξεχάσω κάτι. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ και, καταδικάζω και εγώ ε, ε, αυτή τη φρικαλαιότητα που έλαβε χώρα χθε το Πανεπιστήμιο στο Χαλέπι και σίγουρα συμφωνείτε όλοι μαζί μου. Συμφωνώ και με τον κύριο Σαλαφράγκα σε ό,τι αφορά την, τις ενδεχόμενες καταστροφές ε, ε, περαιτέρω θανάτους και εμβάθυνση της ανθρωπιστικής κρίσης αν συνεχιστεί επαόριστον ε, αυτή η σύγκρουση. Γι' αυτό και πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας. Ε, πιο ειδικά σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για τις συζητήσεις στη Γενέβη και τις τριμερείς συναντήσεις που έλαβαν χώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετείχε. Ήταν η δεύτερη συνάντηση μεταξύ του κυρίου Μπραχήμι ε, τον ΗΠΑ και της Ρωσίας και ήταν ε, στόχος του κυρίου Μπραχήμη να μείνει αυτός ε, ο διάλογος μεταξύ των τριών εταίρων. Όμως εμείς βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και επικοινωνία μαζί του και την ομάδα του και συνεχώς ενημερωνόμαστε σε ό,τι αφορά τη ε, την πρόοδο που έχει σημειωθεί, τις συζητήσεις ε, που διεξάγει και ούτω καθεξής. Και αυτό βεβαίω είναι δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχει με κάθε δυνατό τρόπο όπου υπάρχει δυνατότητα να συμβάλλουμε. Προς απάντηση της κυρία Χίσερ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε σε όλες ε, τις προσπάθειες που αφορούσαν την την ευθύνη και στη Γενέβη και στη Νέα Υόρκη και αυτό θα συνεχιστεί. Η κυρία Σάκ ε, ανέφερε κάποια ζητήματα. Συγγνώμη αν τα προφέρω λάθος τα ονόματά σας. Κάνω ό,τι μπορώ. Η κυρία Φλότρε. Ε, έχουμε όλη επίγνωση των αδυναμιών μας σε ό,τι αφορά τις ε, κοινέ μας προσπάθειες, είτε σε διπλωματικό είτε σε ανθρωπιστικό επίπεδο δεν είναι τέλεια η διαδικασία που ακολουθείται, αυτό είναι σίγουρο. Όμως η κατάσταση, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να απλουστευτεί. Όπως συμβαίνει κάποιες φορές. Πρέπει να εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα, όλες τις πλευρές και όλες τις δυνατότητες ε, για συνεργασία με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως ε, ε, υπέδειξε και η κυρία Γεωργίευα. Συνεργασία λοιπόν με τους ε, επιμέρους φορείς και οργανισμούς ε, για να συμβάλλουμε στο μέγιστο, ούτως ώστε η ανθρωπιστική δράση να πληρώσει του, τους στόχους της, δηλαδή την, τον μετριασμό της ανθρωπιστικής κρίσης. Και βεβαίως και Ξέρουμε πόσο δρυμή ε, είναι ο χειμώνα ε, στη Συρία αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε λοιπόν σε επαφή μαζί με, ε, με αυτούς τους φορείς και οργανώσεις με πολύ συντονισμένο τρόπο και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους βοηθήσουμε επί τόπου. Αυτή η αποφασιστικότητα και η δέσμευσή μα λοιπόν μεταφράζεται και σε έμπρακτη βοήθεια και αυτό θα συνεχιστεί. Συνοψίζοντα θα ήθελα να πω ότι η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ε, οργάνων είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να συνεχιστεί το καθημερινό έργο και οι καθημερινές προσπάθειες ε, και στο ανθρωπιστικό και στο πολιτικό ε, σκηνικό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία έχουμε για να ε, παράσχουμε συνδρομή και στήριξη και προστασία για τους αμάχους. Αυτή είναι η άμεση και πιο πιεστική προτεραιότητα. Θα εστιαστούμε στην εξέβρεση καλύτερων τρόπων για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί θα αναθεωρήσουμε τις ε, κυρώσεις μας ε, στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να μην μεταφερθεί η σύγκρουση σε άλλα, σε άλλα γειτονικά κράτη. Σε αυτό αναφέρθηκαν αρκετά μέλη του Κοινοβουλίου εδώ. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο καθώς και περαιτέρω αποσταθεροποίηση μιας έτσι κι αλλιώς ε, ε, ε, εύκολα μεταβαλλόμενης περιοχής. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε για την παρέμβασή σας. Κλείνει λοιπόν αυτή η συζήτηση. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι κοινή συζήτηση για τη Συμφωνία Τελικής Σχέσης